πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξη. καταρχήν να την εγκρίνουμε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει. θεωρώ ότι εγκρίνεται. Και να εγκρίνουμε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Συμφωνήθηκαν και αυτά. Άρα προχωρούμε προς την ακρόαση και θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι οι συντονιστές θα συνεδριάσουν στο τέλος. Δυνάμει του άρθρου 30 του κανονισμού για την υπηρεσία υποστήριξης για το άσυλο προβλέπεται μία ακρόαση του πρώτου υποψηφίου με τον πρώτο υποψήφιο, μετά από έγκριση στη Βαλέτα από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο επέλεξε τον κύριο Ρόμπερτ Φίσερ από την Ολλανδία. Άρα, θα ακούσουμε τον κύριο Φίσερ. Θα θέλαμε να τον συγχαρούμε καταρχήν για την επιτυχία σε αυτή τη διαδικασία επιλογής και στη συνέχεια θα συζητήσουμε για το πώς θα κινηθούμε στο μέλλον, διότι δυνάμει του άρθρου 30 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου ε, αναφέρεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει για την διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το άσυλο. Θα δούμε κατά πόσο θα γνωμοδοτήσουμε ή όχι. Αυτό θα, γι' αυτό θα αποφανθούν οι συντονιστές μετά. Γι' αυτό και θα διακόψουμε για 10 λεπτά τις εργασίες μας, έτσι ώστε οι συντονιστές να ορίσουν τη θέση τους και στη συνέχεια η Επιτροπή θα, επανεκκινήσει, θα συνεχίσει με τις εργασίες της για να δούμε κατά πώς θα εγκρίνουμε τη θέση των συντονιστών. Μετά από αυτή την υπόδειξη εργασίας θα θέλαμε να ακούσουμε τον κύριο Φίσερ. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να ε, σας υποβάλω την υποψηφιότητά μου ως ε, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ε, Υποστήριξης Ασύλου. Η ΕΑΣΟ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου, είναι μια υπηρεσία που ορίζει μία κοινή ε, πορεία και γραμμή ως προς την πολιτική ασύλου με βάση τις ε, αιτήσει χορήγησης ασύλου, τις οποίες εξετάζει δίκαια και κατά το ταχύτερο δυνατό. Χρειάζεται η ε, δημόσια και πολιτική υποστήριξη για την πολιτική ασύλου. Αυτά είναι θέματα που αφορούν ιδιαίτερα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχουν κοινά πρότυπα και προδιαγραφές κατά την διαχείριση της πολιτικής ασύλου για να ορίσουμε και τις μεταναστευτικές ροές. Σε πολιτικό επίπεδο, το Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισαν για μια πολιτική ασύλου και τους συνεπείς, ε, τις πολιτικές που συνεπάγονται. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε συγκρίσιμη εφαρμογή και ανάλογες πρακτικές με βάση τους κοινού κανονισμούς. Και πώς μπορούμε να εγγυηθούμε τη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις χορήγησης ασύλου η υπηρεσία υποστήριξης χορήγησης ασύλου μπορεί να προβλέψει προς αυτές τις κατευθύνσεις. Η ΕΑΣΟ μπορεί να ορίσει ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου και να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη. Η ΕΑΣΟ θα είναι ένα ανεξάρτητο κέντρο πραγματογνωμοσύνης έτσι ώστε να συντονίσουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στοχεύει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες καθώς και τεχνοοικονομική, τεχνικοηλική υποστήριξη και θα είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που θα λειτουργεί με διαφάνεια μέσα στα πλαίσια της πραγματογνωμοσύνης και της πείρας μας. Η απάντησή μας θα είναι να είμαστε ένα όργανο αλληλεγγύης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θα προσπαθήσουμε να ερχόμαστε σε επαφή και με το Frontex και με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών Υποστήριξης των Προσφύγων. Επίσης, θα συσταθεί ένα συμβουλευτικό φόρουμ προς αυτή την κατεύθυνση. Όλα αυτά αφορούν τη μελλοντική εργασία της ΕΑΣΟ μέσα στα πλαίσια τριών προοπτικών. Από την κοινή πολιτική θα πρέπει να φτάσουμε στην κοινή πρακτική. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε πραγματικές κοινέ πρακτικές, σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση μια κοινή πολιτική. Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε την κοινή εφαρμογή και σύγκληση πρακτικών, εθνικών πρακτικών ασύλου. Η δεύτερη προοπτική είναι από τις βασικές πρακτικές να φτάσουμε στην κοινή πολιτική σε μια κοινή πολιτική. Η ΕΑΣΟ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για νέες πολιτικές και νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις γνώσεις σε μία ε, ανάντη προσέγγιση του θέματος. Η τρίτη προοπτική είναι να μας απασχολήσουν τα κοινά προβλήματα για να φτάσουμε σε κοινέ λύσεις. Πρόκειται για μία οριζόντια προσέγγιση έμπρακτη συνεργασίας με ανταλλαγή απόψεων, κοινή κατάρτιση, κοινέ δράσεις και αποστολές στη στιγμή που υπάρχουν συναφείς αιτήσει. Η εργασία της ΕΑΣΟ έχει διάφορες πτυχές. Καταρχήν μιλάμε για την λειτουργική υποστήριξη για την ανάπτυξη δυνατοτήτων. Σημαίνει ότι υποστηρίζουμε τις εθνικές υπηρεσίες ασύλου με βάση τις αιτήσει που υποβάλλονται για να μπορέσουμε να δώσουμε συμβουλές σε όλους τους τομείς, τους τομείς υγείας, εκπαίδευσης, γλώσσας κλπ σημαίνει και επίγουσα βοήθεια προς κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ε, ιδιαίτερη πίεση στον τομέα του ασύλου. Και επίσης θα υπάρξει ένα κοινό γραφείο ανάλυσης των αιτήσεων των κρατών μελών. Έτσι μπορούν να συσταθούν ομάδες ε, υποστήριξης σε περίπτωση συγκεκριμένων πιέσεων. Ως προς την κατάρτιση και την ποιότητα, θα επεκταθούμε μέσω κατάρτισης και εργαστηρίων, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές, κοινά εγχειρίδια και κοινέ προδιαγραφές. Τρίτον, πληροφορίες και ανάλυση είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της εργασίας. Θα δούμε τις αναλύσεις μέσα στα πλαίσια χορήγησης ασύλου, συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και την ετήσια έκθεση χορήγησης ασύλου. Υπάρχει και η εξωτερική ε, πτυχή για την υποστήριξη τρίτων χωρών. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη ε, δυνατοτήτων και ικανοτήτων σε χώρες ε, υποδοχής, χώρες προέλευσης και χώρες διαμετακόμισης, έτσι ώστε να υπάρχουν διαρκείς λύσεις, να εξευρεθούν διαρκείς λύσεις μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής. Επίσης, έχουμε την συνεργασία του Front Office το οποίο θα μπορούσε να συνδράμει τα κράτη-μέλη και την εργασία των Ηνωμένων Εθνών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΑΣΟ δεν θα είναι το μόνο όργανο υποστήριξης στον τομέα του ασύλου. Θα υπάρχει μια εθελοντική βάση διμερών σχέσεων μεταξύ κρατών μελών, η οποία θα, να, θα συνεχίσει να υφίσταται. Η ΕΑΣΟ δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις σε σχέση με τις μεμονωμένες, μεμονωμένες αιτήσει χορήγησης ασύλου. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τις πρακτικές και λειτουργικές πτυχές στα κράτη-μέλη και τα ίδια τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν επί των αιτήσεων χορήγησης ασύλου. Η ΆΣΟ είναι μια νέα οργάνωση η οποία θα συσταθεί εκ του μηδενός και θα πρέπει να επανδρωθεί. Αλλά δεν θα περιμένω μέχρι τότε έτσι ώστε να αρχίσουμε τις εργασίες μας. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές κατά το πρώτο έτος εργασίας και θα επικεντρωθούμε σε τρία θέματα. Καταρχήν την μεταφορά επιτυχών πιλωτικών προγραμμάτων που έχουν συσταθεί όπως το Eurosil, το ε, European ε, Asylum Curriculum και το Interpreters Pool. Επίσης θα προσπαθήσουμε να διαδώσουμε πληροφορίες στη χώρα προέλευσης μέσω ενός κοινού ιστοτόπου. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα εθνικά σχέδια δράσης. Θα είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι και όταν επανδρωθεί η υπηρεσία μας θα είμαστε ιδιαίτερα δραστήριοι στα, ως προς τα εθνικά σχέδια δράσης. Αυτό αφορά και τη σύσταση μιας υπηρεσίας υποδοχής, κατάρτιση και ποιοτικά σχέδια πείρα των κρατών μελών είναι ζωτική σημασία για την επιτυχία αυτών των προγραμμάτων. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ο κανονισμός της ΕΑΣΟ μιλά για άμεση σχέση και λογοδοσία του Γενικού Διευθυντή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα το προωθήσω αυτό διότι είμαι πεπισμένος για την προστιθέμενη αξία αυτού του οργανισμού στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε αυτή την κοινή εργασία μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής οικοδόμησης μιας κοινή πολιτικής ασύλου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε κύριε Φίσερ. Και ευχαριστώ που υπήρξατε και σύντομος, γιατί έτσι μας διευκολύνεται. να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Όπως είπα λοιπόν και πριν, αρχίζουμε τώρα μια σύντομη συζήτηση. Πρώτα ε, θα λάβουν το λόγο οι συντονιστές, εν προκειμένου ο κύριος Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Φίσερ για την ε, ομιλία σας, συγχαρητήρια για την επιλογή σας. Εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος σας εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας. Το Λαϊκό Κόμμα θεωρεί ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο είναι σημαντικό βήμα για την εκπόνηση μιας κοινή πολιτικής για το άσυλο. Χαίρομαι επίσης που σας άκουσα να αναφέρεστε προς το τέλος της παρεμβάσεώς σας στην υποστήριξη που θα δίνει το ΕΑΣΟ στο εθνικό στο ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσεως, διότι μόλις πριν την προηγούμενη εβδομάδα αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας μετέβη στην Αθήνα και διαπιστώσαμε όμως σώμασιν πόσο μεγάλη βοήθεια χρειάζεται η Ελλάδα για να μπορέσει να διασφαλίσει ώστε η εθνική της διοικητική ικανότητα να είναι αρκετά να είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα επαρκής και αποτελεσματική στην Αθήνα δεν είδαμε να υπάρχει σύστημα αποτελεσματικό. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ρόλος της ΕΑΣΟ θα είναι σημαντικός εν προκειμένου. Τώρα, ερωτήσεις. Τρεις παρακαλώ. Πρώτη αναφέρεται στην αλληλεγγύη, στον μηχανισμό αλληλεγγύης. Δεν αναφερθήκατε ιδιαίτερα σε αυτό στην ομιλία σας κύριε Φίσερ. Γνωρίζετε όμως ότι η παρούσα Επιτροπή αλλά και το παρόν Κοινοβούλιο αναμένουν από την ΕΑΣΟ να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη δηλαδή με τους ανθρώπου που ζητούν άσυλο, αλλά επίσης, και αυτό είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, αλληλεγγύη και με τις χώρες εκείνες μέλη που επί του παρόντος αναλαμβάνουν, επομίζονται το μεγαλύτερο μέρος του βάρου, των αριθμών των προσώπων που ζητούν άσυλο και που εν τέλει προσπαθούν να τα καταφέρουν μόνες τους. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι τι σχέδια έχετε ώστε να διασφαλίσετε ότι η ΕΑΣΟ θα αναπτυχθεί αλλά ότι επίσης θα φροντίσει να εφαρμοστεί ένας επαρκής μηχανισμός αλληλεγγύης. Θυμίζω και το πιλωτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε το 2009 για την Μάλτα ιδίω και ελπίζω να μπορέσει να επεκταθεί και σε άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Είναι σαφές όμως ότι το πιλωτικό κοινό πρόγραμμα δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικό. Δεύτερη ερώτηση. Μη συνοδευόμενοι ανήλικοι. Το θέμα δηλαδή των παιδιών και ιδίω των μη συνοδευόμενων ανήλικων παιδιών που είναι ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα και ανισχύει ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσουμε επί νέα για την σώματεμπορία που περιλαμβάνει και ειδικό άρθρο για τις ανάγκες των παιδιών ανήλικων ε, ασυνόδευτων παιδιών που συχνά είναι μετανάστες που περνούν τα εξωτερικά μας σύνορα και που συχνά επίσης είναι πρόσωπα που ζητούν άσυλο και που είναι οι ομάδες αυτές καθεαυτήν πρόκληση. Άκουσα επίσης να λέτε ότι θέλετε να διατηρήσετε επαφή με, την, με, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς είμαστε η αρμόδια επιτροπή που καθοδηγήσαμε τα βήματα του Κοινοβουλίου χάρη και στην εισηγήτριά μας κυρία Λάμπερτ για την ε, δημιουργία της ε, υπηρεσίας σας και εμείς λοιπόν ενδιαφερόμαστε πολύ να ε, υπάρξει αυτή η διασύνδεση και η επαφή. Πώς βλέπετε ότι μπορεί να γίνει. Ας ακούσουμε πρώτα και τους υπολείπους συντονιστές και θα επανέλθουμε στον υποψήφιο. Και Γκυλιόμ. Καλημέρα σας. Συγγνώμη που καθυστέρησα λίγο στην καθυστέρηση. Συγχαρητήρια κυρία για, την, ε, για τον διορισμό σας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Θα ήθελα όμως ε, να αναφερθώ στις αρμοδιότητες που περιγράψατε ε, τις αρμοδιότητες του γραφείου μεταξύ των οποίων η πιο σημαντική είναι η πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών όπως επίσης η υποστήριξη στα κράτη εκείνα που υπόκεινται σημαντικές πιέσεις. Επίσης, συνεισφορά στην εφαρμογή του κοινού καθεστώτος ασύλου για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων. Εμείς περιμένουμε το γραφείο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακόμη και αν χρειαστεί καιρός για να στηθεί, θα πρέπει οι δραστηριότητες του να ξεκινήσουν το συντομότερο με, τις μελλοντικές σας, με τους μελλοντικούς σας συνεργάτες. Τρεις ερωτήσεις, πολύ σύντομα. Για αυτές λοιπόν τις αρμοδιότητες που περιέγραψα, που, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικές, εσείς ε, τι πιστεύετε, ποιες προτεραιότητες ε, θα δώσετε στις αρμοδιότητές σας, με τι θα ξεκινήσετε όταν ε, αρχίσετε να λειτουργείτε. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς σκοπεύετε να δράσετε εναντί των χωρών των λεγόμενων με ιδιαίτερη πίεση. Και σίγουρα αν το γραφείο δεν είναι πια το α και το ω για την επίλυση όλων των προβλημάτων ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα, το πακέτο ασύλου έχει κολλήσει σε πολλά πακέτα οδηγιώνα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτήν την εναρμόνιση προς τα πάνω, μέχρι πού μπορεί να φτάσει όλη αυτή η εναρμόνιση διαδικασιών. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βίσεφ να σας συγχαρώ για, τον, ε, για την υποψηφιότητά σας, γιατί ο, ο διορισμός σας εξαρτάται από τη διαδικασία έγκρισης που εξαρτάται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Μία αφορά το πολιτικό επίπεδο και άλλη το πολιτικό Θα ήθελα να μας πείτε πότε θεωρείτε ότι θα, είναι, θα καταστεί λειτουργική αυτή η υπηρεσία. Φαντάζομαι θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, ένα έτος, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε θα λειτουργεί πλήρως, πότε θα λειτουργήσει πλήρως αυτή η υπηρεσία. Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η σχέση μεταξύ ΑΣΟ και κρατών μελών σε σχέση με την ανεξαρτησία αυτής της ε, υπηρεσίας. Γιατί δεν είναι ένα θεωρητικό καθαρά ζήτημα, δηλαδή τι πρέπει να κάνετε εσείς, αλλά πώς μπορείτε να διατηρήσετε αυτή την ανεξαρτησία και τι σημαίνει για εσάς. Επίσης, σε πολιτικό επίπεδο, έχει σημασία το πώς θα συνεργαστείτε με άλλους φορείς και οργανισμούς που σχετίζονται με το άσυλο και την πολιτική Frontex. Σε επίπεδο καθαρά διαχείρισης γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διορίσουν τους εμπειρογνώμονες, αλλά εσείς θα είσαστε ο υπεύθυνος αυτής της υπηρεσίας. Πώς θα ε, διαδραματίσετε έναν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να μην γνωρίζετε πώς το προσωπικό σας ε, διευθετεί και επιλύει τα διάφορα ζητήματα. Ευχαριστούμε κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Φίσερ για τον διορισμό σας. Για τους πράσινους η δημιουργία του Γραφείου Ασύλου είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό. Οι ετώντες στο άσυλο θα ξέρουν πια τι θα τους περιμένει. Θα ξεπεράσουμε δηλαδή τη φάση των μεμονωμένων εξετάσεων αιτήσεων, ασύλου από τα κράτη-μέλη. Μετά την επίσκεψη στην Αθήνα, αντελήφθην πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σας διότι στην Αθήνα συναντήσα, συναντήσαμε έναν ε, ε, ετούντα το άσυλο ο οποίος ε, παρά το γεγονός ότι πληρούσε τις συνθήκες του Δουβλίνου απελάθηκε. Σε πολλές χώρες συμβαίνουν τα αντίστοιχα. Ελπίζω λοιπόν ότι σε αυτήν την ανομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας εσείς θα παίξετε το ρόλο σας. Αντιμετωπίζουμε μια κρίση στην Ελλάδα για θέματα ασύλου και ε, μετανάστευσης. Ε, ξέρετε ότι έχουμε φύλακες του Frontex οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα. Θέλω να ξέρω εσείς τι σκέφτεστε σχετικά με την ομάδα υποστήριξης για θέματα ασύλου. Τι σκέφτεστε για τις δυνάμεις πήγουσας παρέμβασης του Frontex. Πώς θα δεσμευτείτε ώστε το Γραφείο Υποστήριξης να σεβαστεί το δικαίωμα ασύλου από ό,τι καταλάβαμε στην Αθήνα, το Frontex δεν είναι ο καταλληλότερος τόπος για να καταθέσει κανείς αίτηση ασύλου. Πού θα πρέπει να κατατίθεται αυτή η πρώτη αίτηση ασύλου, ώστε να μην απορρίπτεται. Και θα ήθελα να μιλήσει και ο συγητής σχετικά. Επειδή δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος από τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Σταβάρες έχει το λόγο από την ΚΟΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Επιτροπή συγκεκριμένα προσδίδει μεγάλη σημασία στις εργασίες ε, για την ΕΑΣΟ. Συμμετείχαμε την Τζιν Λάμπερτ σε αυτή την εργασία συγκρότησης και χαίρομαι που βρίσκεστε τώρα πλέον εδώ και αυτή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία έχει συσταθεί. Ελπίζω να είναι η απαρχή ενός πολύ ε, θετικού διαλόγου μεταξύ μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο μπορείτε να παρίσταστε εδώ όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις και να μας δώσετε πληροφορίες, λεπτομέρειες και τεκμηρίωση ως προς τα ανακύπτοντα ζητήματα. Ως Γενικός Διευθυντής θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τα 500 εκατομμύρια πολίτες μας. Το θέμα του Δουβλίνου ακούσαμε πολλές φορές ότι έχει καταρριφθεί το σύστημα του Δουβλίνου. Θα ήθελα την προσωπική σας άποψη γιατί είναι πολύ καλή ευκαιρία να ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις σας. Θεωρείτε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί αυτό το σύστημα και πώς θα το προωθούσατε αν σας δινόταν η ευκαιρία. Ένα τρίτο ζήτημα αφορά την επανεγκατάσταση. Εγώ συμμετείχα σε μια διαδικασία συναπόφασης σε σχέση με το Ταμείο προσφύγων και ένα ενδεχόμενο πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Αυτά τα δύο προγράμματα ενεκρίθησαν με μεγάλη πλειοψηφία από όλο το πολιτικό φάσμα, από τους συντηρητικούς μέχρι τους κομμουνιστές, γιατί πιστεύουμε στην επανεισδοχή, επανεγκατάσταση των προσφύγων γιατί μιλάμε για 5.000 ετησίως έναντι των 80.000 στις ΙΠΑ και των 200.000 που προβλέπει η τη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Θα πρέπει να υπάρχει μία μόνιμη μονάδα με το κατάλληλο προσωπικό και θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία σωστή υποστήριξη μέσω ΕΑΣΟ ως προς το δικαίωμα επανεγκατάστασης. Θα ήθελα να σας πω πώς θα συσταθεί αυτή η μονάδα επανεγκατάστασης στην ΕΑΣΟ και πώς θα λειτουργήσει, γιατί μιλήσατε για επανεγκατάσταση κατά την παρουσίασή σας και είπατε ότι έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας έμπρακτα για τη σύσταση αυτής της μονάδας. Οι μη εγγεγραμμένοι δεν έχουν πρόθεση να συμμετάσχουν στη συζήτηση, άρα στρεφόμαστε στον κύριο Φίσερ για να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Για 7 λεπτά, έτσι ώστε να έχουμε λίγο χρόνο για άλλα μέλη που θα ήθελαν να παρέμβουν και να έχουμε ένα δεύτερο γύρο ερωταποκρίσεων. Ο κύριος Φίσερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και, τις, και τους αξιωτήμους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Επιτρέψτε μου πρώτα να τονίσω, όπως προσπάθησα να κάνω και στην εισαγωγική μου ομιλία, να τονίσω ότι είμαι πλήρως πεπισμένος ότι η Ευρώπη έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο τρόπο ώστε ένα κοινό ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου είναι πλέον μια ανάγκη. Και για την αναπτυσσόμενη συνεργασία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και λόγω του ότι το θέμα είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα και χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη. Η Ευρώπη έχει και ανθρωπιστικά στάνταρ τα οποία οφείλει να πληρεί. Και για να πληρούνται αυτά χρειάζεται κάποια οργάνωση. όσον αφορά την ΕΑΣΟ μπορεί να παίξει ρόλο και σε ό,τι με αφορά εμένα θα παίξει. Επιτρέψτε μου να ομαδοποιήσω λίγο τις διάφορες ερωτήσεις και να αρχίσω με το θέμα της αλληλεγγύης και του μηχανισμού αλληλεγγύης. Γνωρίζω τις συζητήσεις που διεξάγονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζω και τις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται για το θέμα αυτό. Δεν μπορώ εγώ ωστόσο να αναμειχθώ ως ε, εκπρόσωπος ενός επιχειρησιακού οργανισμού όπως είναι η ΆΣΟ. Η αλληλεγγύη κατά τη γνώμη μου ωστόσο θα πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη. συζητήσει περί οικειοθελούς ή μη χαρακτήρα εκεί δεν μπορεί να αποφασίσει η ΕΑΣΟ. Η ΕΑΣΟ μπορεί να παίξει έναν πρακτικό ρόλο. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα αυτά που συμβαίνουν τώρα μπορεί, μπορούν να προσφέρουν και ευκαιρίες συζητήσεων στο επιχειρησιακό επίπεδο. Εάν δηλαδή μπορεί να δοθεί κάποια αλληλεγγύη και με την έννοια που την εξήγησε ο κ. Μπουσουτήλ Μπορεί λοιπόν να δοθεί και στην ειδική αυτή περίπτωση. Υπάρχουν ενδεχομένω πολλέ απαντήσει που πρέπει να δοθούν στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κατάσταση στην Ελλάδα. Να αρχίσει τώρα η ΕΑΣΟ να συζητεί την πρακτική πλευρά, αυτό μπορεί να συμβάλλει σε μια ευρύτερη ε, συζήτηση περί Το θέμα της επανεγκατάστασης που συνδέεται στενά. Διάβασα βέβαια την έκθεση, σημαντική έκθεση, που περιέχει και πολλές πρακτικές προτάσεις. Εδώ μπορώ να πω λίγο αυτά που είπα και προηγουμένως. Γνωρίζω την πολιτική συζήτηση που διεξάγεται και θεωρώ ότι και εδώ δεν θα ήταν σκόπιμο ένας οργανισμός να προσπαθήσει να αναμειχθεί σε μια πολιτική συζήτηση. Ταυτόχρονα η επαναγκατάσταση που αποτελεί και μακρά παράδοση στην χώρα από την οποία προέρχομαι είναι μία από τις λύσεις στον τομέα της μετανάστευσης με την κατάσταση και ανακατανομή είναι πράγματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν. Όπως είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία, η ΕΑΣΟ ασφαλώς θα είναι διαθέσιμη να αναλάβει ρόλο στο θέμα αυτό και στην εξωτερική και στην εσωτερική επανεγκατάσταση. Θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο πρώτου βαθμού. Και βεβαίως και οι χώρες μέλη αλλά και ο ύπατος αρμοστή για του πρόσφυγες των ΗΕ έχουν ρόλο να παίξουν, αλλά και ΑΣΟ μπορεί να παίξει ρόλο και ελπίζω μάλιστα που τέτοιο ρόλο που θα προσφέρει και ιδέε και κίνητρα, γιατί το θέμα είναι βέβαια θέμα που προκαλεί ανησυχίε και όσο μπορεί να παίξει ρόλο η ΑΣΟ θα παίξει. περί ασυνόδευτων ανηλίκων τώρα. Όπως είπε ο κύριος Μπουσουτήλ προηγουμένως, το θέμα είναι πολύ ευρύτερο ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα γραφείο ασύλου από μόνο του. Από την άλλη μεριά είναι και μια από τις σημαντικές τάσεις που διαπιστώνονται στις μεταναστευτικές ροές. Μέρος λοιπόν του έργου του ΕΑΣΟ θα είναι και στην πλευρά της εκπαίδευσης αρχικά να εξεταστούν και να πρόχθουν γιατί οι τρόποι που αντιμετωπίζονται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ διαφορετικοί. Για παράδειγμα, πληροφορίες που παρέχουν οι χώρες προέλευσης η ΕΑΣΟ μπορεί να παίξει ένα ρόλο ώστε να καταστούν πιο ορατές και πιο απτές οι διαστάσεις του προβλήματος. Σχετικά τώρα με τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες. Μία προτεραιότητα είναι δεδομένη το ελληνικό εθνικό σχέδιο δράσεως ήδη πριν από την δημιουργία του ΕΑΣΟ. Θα βρίσκεται λοιπόν επικεφαλής της λίστας των προτεραιοτήτων μας. Το δεύτερο το έχει ήδη κρίνει ο κανονισμός, ότι ο αριθμός δηλαδή project που έχουν ήδη αρχίσει θα πρέπει να αναλυθούν από την νέα οργάνωση και μάλιστα με τρόπο ομαλό. Ε, πρόκειται για ε, προγράμματα, για project τα οποία ήδη κινούνται και αποδίδουν. Επίσης ένα από τα σημαντικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν εξ αρχής είναι να επεξεργαστούμε αυτή την αρχή της πληροφορίας των πληροφοριών που δίνουν χώρες προελεύσεως. Εδώ μια ευρωπαϊκή προσέγγιση μπορεί να αποδώσει προστιθέμενη αξία για προφανείς λόγους. Για λιγότερο προφανείς λόγους, αλλά ίσως και κανένα φορά για προφανείς λόγους, ορισμένες χώρες το φοβούνται αυτό. Εδώ διεξάγεται πολλή συζήτηση σχετικά με τις πληροφορίες της χώρας προέλευσης και νομίζω πάντως ότι υπάρχουν πράγματα να, από εδώ, να κερδιθούν από εδώ. Λόγω του μεγέθους του οργανισμού δεν θα ήταν νομίζω σκόπιμο για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του να αποφασιστούν περισσότερες προτεραιότητες από αυτές. Και πάντως αυτό δεν πρόκειται, θα κρυθεί εδώ μάλλον και όχι ε, σε εμά. Τώρα, οι ορισμοί που περιλαμβάνει ο κανονισμός είναι σωστοί. Αναμένω και αυτό νομίζω είναι το νόημα της ερώτησης αναμένω ότι θα αναπτυχθούν συζητήσεις σε κάθε δεδομένη στιγμή. Οι λύσεις θα πρέπει να είναι βέβαια τέτοιες που να αντιμετωπίζουν τις πιέσεις. Να δοθεί τώρα ορισμός αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι είναι δικό μου καθήκον για αρμοδιότητα. Οι προσδοκίες, καθώς επίσης πότε θα είναι λειτουργικό το γραφείο, ένα μέρος το αποφασίσατε εσείς, διότι περιλαμβάνεται στον κανονισμό 19 Ιουνίου, του επόμενο έτους, 19 Έκτου, θα πρέπει ε, να είναι έτοιμο και λειτουργικό, επιχειρησιακό ε, το γραφείο. Αυτό το καθήκον μας έχετε αναθέσει και θα αποκριθούμε. Μέσα στην διάρκεια του επόμενου έτους προβλέπω να είναι επιχειρησιακό το γραφείο. Αλλά ήδη πριν από αυτό και λόγω των αντικειμένων που ανέφερα πριν, ελπίζω ότι θα έχουμε ήδη επαρκές προσωπικό που θα είναι ε, ήδη έτοιμο να αρχίσει να εργάζεται και θα περιμένουμε απαραίτητα τον Ιούνιο. Ε, η ερώτηση σχετικά με την κατάσταση. Εδώ νομίζω καθίσταται ανάγλυφη η δυνατότητα προσφοράς προσθέμενης αξίας από την ΕΑΣΟ στον κανονισμό του Δουβλίνου αναφέρεται η πραγματογνωμοσύνη και η γνώση και επιχειρησιακή και ε, επί του πεδίου Νομίζω αυτό το ανέμενε και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι το ΕΑΣΟ θα μπορέσει να το καταστήσει αυτό σαφές και θα μπορέσει να επιλύσει τα πρακτικά αυτά προβλήματα. Ε, άλλη ερώτηση τώρα για την Ελλάδα και το Frontex. Υπάρχει διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ Frontex και ΕΑΣΟ. Αλλά υπάρχουν και μίσο που θα πρέπει να συνεργάζονται στενά οι δύο φορείς. Στο σχέδιο δράσεως της Κομισιόν Ήδη διαλαμβάνεται αυτό ότι η ΑΣΟ θα πρέπει να αρχίσει πολύ σύντομα να σκέπτεται πώς θα εκπαιδεύει τα πρόσωπα που εργάζονται για το Frontex, είτε είναι εμπειρογνώμονες είτε είναι μεθοριακοί φρουροί για την αντιμετώπιση ανθρώπων που προσέρχονται και ζητούν άσυλο και έχουν το δικαίωμα να το πράξουν. Εκπαίδευση λοιπόν ασφαλώς θα παίξει ρόλο. Θα είναι σημαντικό στοιχείο δηλαδή στις σχέσεις με την Frontex. Δεύτερο, το σχέδιο δράσεως για την Ελλάδα έχει δύο σκέλη, αφενός τα σύνορα, Frontex επομένως, αφετέρου το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα, που θα είναι ο βασικός στόχος του ΕΑΣΟ. για το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο δεν έχει καταρρεύσει κατά την δική μου επαγγελματική άποψη. Εν μέρη ίσως. Η σχέση με την Ελλάδα, ναι, ε, έχει χαλάσει, αλλά όχι με τις άλλες χώρες και εφόσον δεν έχουμε τίποτε καλύτερο από το σύστημα αυτό, καλύτερα να προσπαθήσουμε να το επισκευάσουμε. Τέλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι ασφαλώς διαθέσιμος για διάλογο και για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας, τεκμηριώσεως ή οτιδήποτε άλλο ε, χρειαστεί η Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε κύριε Φίσερ. Θα ήθελα οι βουλευτές που θα λάβουν το λόγο να τον λάβουν σύντομα έτσι ώστε να τα καταφέρουμε. Η κυρία Χολμάιρ, δύο λεπτά έκαστος παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις. Στην Ελλάδα σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα επιθυμεί να φτιάξει αποκεντρωμένους καταβλισμούς προσφύγων ώστε να αποφύγει, να αποτρέψει την μεγάλη μαζική συγκέντρωσή τους στην Αθήνα και να απαλύνει έτσι και τα προβλήματα. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε την ελληνική αυτή προσπάθεια και στην καταχώρηση και στην επιτάχυνση των διαδικασιών, καταχώρηση δηλαδή, των προσώπων. Δεύτερη ερώτηση. Υπάρχει το ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα του ότι το 95% των προσερχομένων δεν ζητούν άσυλο, αλλά λένε καθαρά και ειλικρινά ότι θέλουν απλώ να περάσουν στην Ευρώπη για λόγου φτώχεια, διότι δεν περνάνε καλά τέλο πάντων στην χώρα τους και δεν βλέπουν να υπάρχουν μελλοντικέ προοπτικές. Θέλουν λοιπόν καλύτερες δυνατότητες κοινωνικές, ευημερίας κλπ. στι χώρε μέλη τι δυνατότητες βλέπετε τώρα για επανεισδοχή, επανεγκατάσταση να βοηθήσετε, να συνδράμετε την Ελλάδα και αυτό ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα που ανεφήσαν από τις συζήτηση με τις ελληνικές αρχές ότι δηλαδή το ποσοστό επανεισδοχής ε, είναι ελάχιστο διότι οι πρεσβείες δεν δέχονται να συνεργαστούν. Άρα ο διάλογος με τις πρεσβείες θα ήταν σημαντικό και βεβαίω θα σας υποστηρίξει η Ευρώπη των 27. δύο λεπτά Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας, κύριε Φίσερ. Συγχαρητήρια. Εγώ τώρα θα ρωτήσω αγγλικά πώς λαμβάνεται υπόψη το πλαίσιο προστασίας με βάση τη σύμβαση της ε, Γενέβης, πώς ορίζεται το στάτους ε, των προσφύγων με βάση ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, τις ε, γυναίκες και τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο. Επίσης, ως προς την ισότητα των δύο φύλων, θεωρούμε ότι η ΕΑΣΟ θα προβάλλει κατάρτιση ε, με βάση τις ανάγκες των φίλων πώς μπορεί η ΕΑΣΟ να συνεισφέρει έτσι ώστε να τηρηθεί η εφαρμογή. Ως προς τις ε, αρχές της ΥΠΑ της αρμοστίας έτσι ώστε να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ των δύο φύλων και πώς λαμβάνεται υπόψη ο, πώς θα αντιμετωπιστεί ο ακροτηριασμός των γεννητικών οργάνων της γυναίκας και πώς η ΕΑΣΟ θα προωθήσει μία πραγματογνωμοσύνη με βάση τις ανάγκες των γυναικών και των ευπαθών ομάδων με βάση τη χώρα προέλευσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομη. Θα σας συγχαρώ κι εγώ για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θέλετε να συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο. Να σας ρωτήσω όμως σύντομα κάτι πιο πολιτικό. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι θέλετε να είστε τίμιος και ουδέτερος. Συμφωνώ. Αλλά σε αυτόν τον τομέα η ουδετερότητα δεν αποτελεί πολυτέλεια, μία πολυτέλεια που δεν μπορείτε να την επιτρέψετε στον εαυτό σας ε, άμα δείτε το κλίμα το οποίο βασιλεύει στις διάφορες χώρες έναντι όλων αυτών των ανθρώπων που για διάφορους λόγους έρχονται στην Ευρώπη και που τα κράτη-μέλη δεν σέβονται τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, ε, Τι θα κάνετε εσείς έναντι των χωρών εκείνων που δεν έχουν καμία πρόθεση να στεβαστούν τους ελάχιστους κανόνες σεβασμού του ασύλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι η επικεφαλής αντιπροσωπείας ε, Λίμπε στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα και σας ευχαριστώ που συνεργάζεστε τόσο ε, ε, ε, ε, τόσο καλά και ευχαριστώ και την γραμματεία επίσης που μας επέτρεψε να πάμε στην Ελλάδα και ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούσαμε και είδαμε. Το σύστημα πλέον έχει μπλοκάρει και υπάρχει μια κοινωνική αντίδραση όλο ένα μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Εγώ θα μιλούσα για κοινωνικο-ανθρωπιστική κρίση Υπάρχουν νομοσχέδια που θα πρέπει να ψηφιστούν τον Ιανουάριο. Είδαν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Κομισιόν. Είδαμε μια, ένα προεδρικό διάταγμα. Άλλα κράτη-μέλη προσφέρουν βοήθεια. Αλλά εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε και συμφώνησε όλη η αντιπροσωπεία είναι ότι η μεταβατική περίοδος η οποία θα αποφασιστεί να παραταθεί για ένα χρόνο. σαν να υπήρχε δηλαδή ένα κενό για αυτές τις 50.000 που εξετάστηκαν. Λοιπόν, το γραφείο τι όθηση μπορεί να δώσει για να γίνει ότι είναι απαραίτητο. Μπορεί να διαθέσει υποδομή. Και Αυτή η μελλοντική ανθρωπιστική κρίση η οποία θα πλήξει την Αθήνα και όχι μόνο την Αθήνα αλλά και άλλες πρωτεύουσες Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, ποιος θα είναι ο ρόλος αυτού του γραφείου, τόσο ώστε να εξωθήσει τα κράτη-μέλη, να λύσουν αυτές τις αντιμαχόμενες καταστάσεις οι οποίες όπου να είναι θα εκραγούν. Κύριε Φίσερ. Νομίζω ότι θα πρέπει να μας βοηθήσετε και εσείς να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια εργασίας. Θα ήθελα να απαντήσετε λοιπόν σε πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις ε, προέκυψαν για την Ελλάδα, το πρόγραμμα δράσης δηλαδή που γνωρίζετε. Κύριε Λάμπερτ, ζητήσατε το λόγο, είχατε στήσει το λόγο, με συγχωρείτε. Η κυρία Λάμπερτ, δεν σας είχα δει. Σας δίνω το λόγο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εγώ ήμουν η συγγήτρια για την ΕΑΣΟ και είχαμε πολύ καλή συνεργασία με όλες τις άλλες πολιτικές ομάδες. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ και που ξεκινούν οι εργασίες της ΕΑΣΟ, διότι θέλουμε να υπάρχει ευρωπαϊκή προσέγγιση και όχι η διακυβερνητική. Γι' αυτό είμαστε υπέρ του, της υπηρεσίας υποστήριξης. Μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας υποστήριξης έγινε λόγος για επιπρόσθετη πραγματογνωμοσύνη και input από την κοινωνία των πολιτών, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς, μη κυβερνητικέ ή τοπικές αρχές που πολλές φορές μας δίνουν επιτόπιες λύσεις. Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας θα πρέπει να προβείτε στη σύσταση της υπηρεσίας κάθε αυτής, Πώς βλέπετε το χρονοδιάγραμμα και πώς αυτό το συμβουλευτικό φόρουμ μπορεί να αποτελέσει προσθέμενη αξία στην εργασία της ΕΑΣΟ. Κύριε Φίσερ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ως προς την Ελλάδα, γνωρίζετε το πρόγραμμα δράσης και τα διάφορα στάδια του η ΕΑΣΟ θα πρέπει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και ως προς την υπηρεσία μετανάστευσης στην Ελλάδα, την οικοδόμησή της, έχει μεγάλη σημασία η κατάρτιση ε, ποιοτικά έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε γενικότερα για να απαντήσω στον ε, διπλανό μου εδώ που με ρώτησε πώς ε, μπορούμε να συνεισφέρουμε. Δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ ΕΑΣΟ, θα πρέπει να είμαστε ένα ανεξάρτητο σώμα και αυτό εξαρτάται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι θα πρέπει να εξισορροπήσουμε όλες τις συνιστώσεις Υπάρχει το λειτουργικό και πολιτικό σκέλος σε κάθε κράτος μέλος. Υπάρχει η Επιτροπή, το κοινό, η κοινωνία των πολιτών, η Πατιαρμοστία. Υπάρχουν τόσοι φορείς που ελπίζω να είμαι αμερόληπτος συνολικά. Αλλά αυτή θα είναι και η πρόκληση. Ως προς την αναγνώριση του ρόλου των δύο φίλων, έχει σημασία, έχουν σημασία οι πληροφορίες από τη χώρα προέλευσης. Γι' αυτό θα πρέπει να συλλέξουμε τις πληροφορίες και εκεί ακριβώς θα πρέπει να γνωστοποιούνται σε αυτό το επίπεδο. Άρα όλα αυτά συνάγονται από τις πληροφορίες από τη χώρα προέλευσης. Και αυτό αφορά και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εάν καταφέρουμε να έχουμε ε, ενίες προδιαγραφές ως προς την ποιότητα και την ουσία σε σχέση και με το ρόλο των δύο φίλων, βεβαίως θα έχουμε όλα τα δεδομένα για να μπορούμε να απαντήσουμε. Για την κοινωνία των πολιτών και το συμβουλευτικό φόρουμ Εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι στο δεύτερο ήμιση του επόμενου έτους θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις εργασίες του το Συμβουλευτικό Φόρουμ, θα ήθελα να δούμε ποιες είναι οι διαφορετικές εμπειρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα συμβουλευτικά φόρουμ και ποιος ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών. Δεν έχω φτάσει σε ένα τελικό συμπέρασμα, αλλά αν κρίνω από την επαγγελματική μου πείρα, η κοινωνία των πολιτών μας δίνει πολλές πληροφορίες ως προς τη συγκρότηση αυτής της πολιτικής και λειτουργικής διαδικασίας και θα σταθώ, θα βασιστώ σε αυτή την πείρα. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Φίσερ για τις απαντήσεις σας. Και όπως είπαμε πριν, τώρα θα διακόψουμε για ένα τέταρτο περίπου, ώστε να μπορέσουν οι συντονιστές να διαμορφώσουν άποψη. Παρακαλώ όλοι στην αίθουσα. Να μας επιτρέψετε να διεξαγάγουμε αυτή τη ε, ε, συνάντηση των συντονιστών. Δέκα λεπτά μας φτάνουν. Καλά, δέκα λεπτά. Για να μην παρατείνουμε πολύ. Προτείνω, συνεχίζει ο Πρόεδρος, να πούμε 15 λεπτά και μετά θα επαναλάβουμε τις ε, εργασίες μας και ε, θα αναλάβει το υπόλοιπο της Επιτροπής να εγκρίνει όχι την πρόταση των συντονιστών.